για το να αυξηθεί η σημασία εμπορίου μεταξύ λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλαβα έξι προτάσει ψηφίσματο για την παράτωση αυτή τη συζήτηση. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαρθεί αύριο στι 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία. Περνάμε στο ζήτημα της Ισλανδίας. Δίνω ένα λεπτό στο Συμβούλιο. Is this a request for catch the eye? Είναι έτοιμα για τη διαδικασία catch the eye. Πολύ ωραία. Okay. Uh, Όπως σας είπα, περνάμε στο θέμα της Ισλανδίας. Έκθεση προόδου 2010. Εξ του Συμβουλίου, η κυρία Γκιόρη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές την, τον θετικό ρόλο που ε, διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον βλέπω, βλέπω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε σχέση και με τις διαπραγματεύσεις αλλά και για τις διαπραγματεύσεις για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι μία από τις πιο σημαντικές ε, εξελίξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομόφωνα αποφάσισε το Συμβούλιο η Ισλανδία να πάρει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Έγινε στις 27 Ιουλίου 2010 μια πρώτη τέτοια συνάντηση και το Νοέμβριο 2010 ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης. Όλα βαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο. Η επόμενη σύνοδος προβλέπεται στις 27 Ιουνίου για το θέμα της Ισλανδίας. Θα έχουμε έτσι την ευκαιρία τα επιτεύγματα, τα αποτελέσματα να επανεξεταστούν προσεκτικά και ελπίζουμε το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια θα μπορέσουν να ανοίξουν. Υπάρχουν σημαντικά θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα και που θέλω ξεχωριστά να τα δούμε. Και το σχέδιο αναφέρει αυτές τις σημαντικές πτυχές. Στην έκθεση προόδου λοιπόν διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι τα πολιτικά κριτήρια τα οποία υλοποιούνται από πλευρά τη χώρα αυτή για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλη την οικονομική κρίση που έπληξε ιδιαίτερα αυτή τη χώρα, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να προετοιμαστεί η Ισλανδία με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα αιτήματα τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δεκέμβριο 2010 τόνισε το Συμβούλιο ότι η δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί εξαιρετικά στην ε, Ισλανδία έχει ισχυρού θεσμού και στενέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η χώρα. Διαπιστώνει περαιτέρω το Συμβούλιο ότι η χώρα αυτή είναι σε θέση να αφομοιώσει, να αποδεχθεί το, το κοινοτικό κεκτημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό και έτσι ε, είναι ήδη όλας μέλος ε, του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Η χώρα λοιπόν αυτή θα πρέπει να επανακτήσει την ικανότητά της ε, να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει επιπλέον στο ότι στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η Ισλανδία να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αφομοιώσει πλήρως ε, τα ευρωπαϊκά κεκτημένα. Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων θα καθοριστεί από το βαθμό και το μέτρο του κατά πόσον θα μπορέσει να υλοποιήσει η Ισλανδία τις απαιτήσει, του όρους και τις προϋποθέσεις σε σχέση με το Συμβούλιο 17 Ιουνίου 2010 και πώς θα λάβει υπόψη τα, ε, τις απαιτήσει ε, που διατυπώνονται και τις ανάγκες που υπάρχουν να καλυφθούν συγκεκριμένοι στόχοι η βάση των, ε, της συνθήκης που καθορίζει την ε, σχέση Ισλανδίας ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το παρελθόν ήταν πολύ δημιουργικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον χώρο Σέγγεν η Ισλανδία. Μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και ενεθάρρυνε την Ισλανδία να προχωρήσει σε αυτή την πορεία. Η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρωμένη εικόνα για τα επιτεύγματα, για τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και τα όσα απομένουν να γίνουν. Έχουμε κοινή δέσμευση, κοινή υποχρέωση. Πρέπει και έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και έναντι των πολιτών τη Ισλανδία να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο ειλικρίνεια και αμεσότητα. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφέ ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα κατά τη διάρκεια τη Ουγγρική Προεδρία. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτό το εγχείρημα βασιζόμαστε στην υποστήριξη όλων των κρατών τη Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει η προώθηση αυτών, ο ρυθμό και ε, η προώθηση αυτών των προσπαθειών να συνεχιστούν κατά του επόμενου μήνε ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία διεύρυνσης. έχω ε, πιστεί ακράδαντα ότι μπορεί να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα και ότι η ένταξη αυτή τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει περαιτέρω έμφαση και θα τονώσει ιδιαίτερα τη διαδικασία διεύρυνση. Χρειαζόμαστε μια ενωμένη, ολοκληρωμένη Ευρώπη. Και αυτό θα είναι μια σημαντική συνεισφορά. Ευχαριστώ. Εξ τη Επιτροπή, ο Επίτροπο ο Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συζήτηση για την Ισλανδία και τα επόμενα βήματα στην προσχώρησή της ε, σήμερα έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη για την προσχώρηση της Ισλανδίας και να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Πρέντα για την πολύ καλή έκθεσή του. Η, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλαν πολύ σημαντικά στην όλη διαδικασία. Εστάλησαν τα σωστά μηνύματα στην Ισλανδία τη σωστή στιγμή. Η αξιολόγηση τη συμμόρφωση τη Ισλανδία με το κοινοτικό κεκτημένο, η διαδικασία ενδελεχού εξέταση έχει ήδη ξεκινήσει. Από τον Νοέμβριο του 2010, 24 24 κεφάλαια έχουν συζητηθεί και 23 23 ενδελεχού εξέταση εξέταση έχουν ολοκληρωθεί συμπεριλαμβανομένων τη γεωργία τη αλληλεία, του περιβάλλοντο, τη περιφερειακή πολιτική και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η διαδικασία τη ενδελεχού εξέταση είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα τεχνική και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων καταφέραμε να εντοπίσουμε ευαίσθητα ζητήματα και προκλήσει. Σε κάποια σημαντικά κεφάλαια, όπω η γεωργία, το περιβάλλον και η αλληλεία. Το στάδιο αυτό λοιπόν της διαδικασίας διαπραγματεύσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ε, περιμένουμε οι διαπραγματεύσεις αυτές καθ' αυτές να ξεκινήσουν προς τα τέλη της Ουγγρικής Προεδρίας, ανοίγοντας κάποια κεφάλαια στις 27 Ιουνίου, τότε τουλάχιστον προβλέπεται. Θεωρώ ότι είναι φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα αυτό και θα επιτρέψει σε όλες τις πλευρές να σημειώσουν πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να καταγράψει την ιδιαιτερότητα και τις προσδοκίες της Ισλανδίας και θέλουμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων να διαφυλάξουμε τις αρχές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, στοχεύουμε να εργαστούμε με τρόπο επικδομητικό και ανοιχτό προκειμένου να καταφέρουμε να βρούμε αποδεκτές λύσεις και για τις δύο πλευρές έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται το υψηλό επίπεδο συνεργασίας το οποίο υφίσταται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ισλανδικών αρχών. Όπως με οποιαδήποτε προσχώρηση, όπως έχει γίνει δηλαδή και στο παρελθόν, δεν αναμένουμε ότι το εγχείρημα θα είναι εύκολο αλλά με την Ισλανδία έχουμε καλύψει ήδη ένα πολύ σημαντικό έδαφος στο δρόμο προς την προσχώρηση. Όπως άλλωστε έχει υποθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως λέτε και εσείς στο ψήφισμά σας, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει ότι το ζήτημα του ICE-SAVE θα επιληθεί γρήγορα. Όσον αφορά τώρα την δημοσιονομική εξυγίανση και ιδίω την εξυγίανση του τραπεζικού τομέα στην ε, Ισλανδία με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκεί τα αποτελέσματα ήταν ε, ε, εντυπωσιακά είναι δεσμευμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει περισσότερο με το θέμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, να αναδιαρθρώσει το χρέος και να ενδυναμώσει την οικονομία της χώρας. Επίσης, η κυβέρνηση εκπονεί μια στρατηγική προκειμένου σιγά-σιγά να πάυσουν οι έλεγχοι για τα κεφάλαια και αυτό θα βοηθήσει να δημιουργηθεί ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στο μέσο προεταγξιακής υποστήριξης μέτρα τα οποία εμείς εφαρμόζουμε. 28 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για τα επόμενα τρία χρόνια προκειμένου να ενδυναμωθεί η δημοσιονομική ικανότητα της Ισλανδίας και να προετοιμαστεί η χώρα αυτή για την διαχείριση των διαφορετικών ταμείων. Επίσης έχει σημειωθεί πολύ καλή πρόοδος στην εκπόνηση των προγραμμάτων για το 2011 και για συγκεκριμένα επιμέρους προγράμματα. Δραστηριότητες επίσης έχουν ξεκινήσει και για τα φορολογικά προγράμματα. Συμφωνώ μαζί σας ότι όντως θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση δημόσια για την προσχώρηση της Ισλανδίας. Νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις πλευρές να εκφράσουν άποψή τους, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την πραγματικότητα, τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα διασκεδάσει οποιοδήποτε ούτε μύθους μπορεί να υπάρχουν και χαιρετίζει το γεγονό ότι ε, οι Ισλανδικέ Αρχέ έχουν ήδη ξεκινήσει μια έντονη διαδικασία ενημέρωση και πληροφόρηση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχει βελτιωθεί η κοινή γνώμη στην Ισλανδία υπέρ τη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω αυτό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτου. Αυτό υποστηρίζει και την όλη διαδικασία προσχώρηση και έχει αλλάξει γενικότερα και η στάση των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αλλάξει και η εικόνα που έχουν οι πολίτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να διαχείσει οποιασδήποτε πληροφορίε απαιτούνται προκειμένου να εμπλουτιστεί όλη η συζήτηση που θα λάβει χώρα. Η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ρέικεβικ συμμετέχει έντονα σε όλε αυτέ τις δραστηριότητε και έχει, θα δημιουργηθεί και ένα νέο κέντρο πληροφόρηση και ενημέρωση Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, προσβλέπω ειλικρινά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδελέχους εξέτασης και στο επίσημο άνοιγμα των κεφαλαίων των διαπραγματευτικών. Ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ε, για 1,5 λεπτό για το Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω ε, την ε, Κομισιόν για το Συμβούλιο και να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα με τα δύο θεσμικά όργανα και για τη σύνταξη αυτού του ψηφίσματος. Όπως είπαμε ε, πριν από 9 μήνες όταν εκφράσαμε τη γνώμη μας για την ε, αίτηση ένταξης της Ισλανδίας ε, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε πρώτα απ' όλα στα πολιτικά κριτήρια. Όντως έχει εξαιρετική παράδοση δημοκρατική η Ισλανδία. Επίσης εκτιμήσαμε την πρόοδο που πραγματοποίησε η χώρα αυτή τους τελευταίους μήνες στην ενίσχυση της ε, του δικαστικού ε, κλάδου ε, σχετικά με τον διορισμό και την ανεξαρτησία των δικαστών. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό τα μέτρα αυτά να υλοποιηθούν στην πράξη. Δεύτερον, τα οικονομικά κριτήρια. Σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Ισλανδία πληρεί πολλά από τα κριτηρία για ένα νέο κράτος μέλος. Και είναι πολύ θετικό ότι αλλάζει η τάση της κοινή γνώμης και ε, φαίνεται ότι όταν θα γίνει το δημοψήφισμα θα τελειώσει αυτή η διαμάχη σχετικά με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θετικό τρόπο. Η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσει την παρουσία της Ευρωπαϊκή Ένωση στην ακτική περιοχή γενικά και στο Αρκτικό Συμβούλιο πιο ειδικά. Ε, είναι απαραίτητο λοιπόν να επιτύχουν οι διαδικασίες αυτές και οι διαπραγματεύσεις ένταξης και γι' αυτό θα πρέπει οι Ισλανδικέ αρχές να ανοίξουν ένα δημόσιο διάλογο με τη συμμετοχή όλων, ε, διότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι δημοσκοπήσει τη κοινή γνώμη δείχνουν ε, βελτίωση τη κοινή γνώμη υπέρ τη ένταξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αυριανή ψηφοφορία είναι ένα από τα στάδια που θα ε, φέρουν πολύ ε, γρήγορα ε, την Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε ο κύριος Πρέντα, η Ισλανδία πραγματοποιεί σημαντικά βήματα πρόοδου, παραδείγματο χάρη είναι ενίσχυση τη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια ειδική επιτροπή που ανέλαβε να ερευνήσει και να αναλύσει τις διαδικασίες που οδήγησαν στην κατάρρευση του του Ισλανδικού τραπεζικού συστήματος, η δημιουργία μιας κοινοβουλευτικής, μικτής κοινοβουλευτικής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλανδίας, η θέση σχετικά με την είσοδο στην ζώνη του ευρώ, η αυξανόμενη εμπειρία ε, που υπάρχει στον ε, ε, τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Το ακαθόδες θέμα του iSafe. Το επόμενο Σάββατο θα γίνει το δημοψήφισμα όπου οι Ισλανδοί θα αποφαθούν με την ψήφο τους. Πέραν αυτού, ε, αυτή η, συζήτηση δείχνει ε, πόσο, ε, πόσο βαθιές είναι οι δημοκρατικές ε, αρχές στη χώρα αυτή, διότι ο λαός της Ισλανδίας συμμετέχει σε αυτή την πολύ λεπτή και ευαίσθητη φάση των διαπραγματεύσεων. Αν δεν έχει θετική έκβαση το δημοψήφισμα, η Ισλανδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε, δημιουργώντας μια οριζόντια ε, δομή και η Ισλανδία έχει δεσμευτεί να αποσμιώσει την Αγγλία και την ε, Ολλανδία για τις ζημιές που έχουν ε, υποστεί. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ασχίσει επιπλέον πιέσεις που θα δημιουργούσαν μια αντίδραση κλεισίματος και αυτοάμυνας εκ μέρους της Ισλανδικής κοινωνίας. Όσον αφορά την Αλία και τη Γεωργία, πιστεύω ότι η Ισλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρουν τις καλύτερες λύσεις για να γίνουν σεβαστά τα κριτήρια κριτήρια της συνθήκης και για να ε, ε, προστατευθεί η Ισλανδική οικονομία, τα οικοσυστήματα και οι ιδιαιτερότητες της χώρας. Η ένταξη της ε, Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σημάνει για την Ευρώπη ότι θα φτάσει μέχρι τα όρια του Βορείου Πόλου με πολύ σημαντικές θετικές συνέπειες από άποψη πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντική και επιστημονική. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη έτσι μετά από 60 χρόνια αποδεικνύει ότι έχει ακόμα μια πολύ, ασκεί ακόμα μια πολύ μεγάλη έλξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το screening process, η διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο, θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η Ισλανδία ως μέλος της του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έχει ήδη εγκρίνει ένα πολύ σημαντικό τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Και από ό,τι φαίνεται το 65% των Ισλανδών θέλουν να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την θέση μου ως επικεφαλής της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προκειμένου να πείσω τους Ισλανδούς να μην οχυρωθούν αυτή τη στιγμή σε ευρωσκεπτικιστικές θέσεις αλλά να αναμένουν την ε, συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Στο Ρέκεβικ θα λάβει χώρα στις 26 και 27 του μηνός η συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, μιας επιτροπής που δημιουργήθηκε για την καλύτερη συζήτηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, του Ισλανδικού Κοινοβουλίου. Λυπάμαι που ε, στις αρχές Μαρτίου δεν καταφέραμε όμως να καταλήξουμε σε μία συμφωνία και ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το, του, το ζήτημα του σκουμπριού των ποσοστώσεων που προβλέπονται δηλαδή από την Ισλανδία ενώ υπάρχουν ήδη επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που λένε ότι η ποσόστοση της Ισλανδίας πρέπει να μειωθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία μικρή χώρα πάντοτε προκαλεί μεγάλους πονοκεφάλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θέλει να γίνει μέλος. Και ξέρουμε τους πονοκεφάλους της Ισλανδίας, το περιβάλλον, την ε, αλία, αλλά έχουμε μια συνταγή για τα προβλήματα αυτά. Είναι ε, μια ε, στάση ανοιχτή, ε, καλωσορίσματος. Πρέπει να, ε, να, να με το μαλακό μια μικρή χώρα. Άκουσα αυτά που υπόθηκαν για το θέμα του κοινοτικού κεκτημένου και του τι κάνει η Ισλανδία γι' αυτό. Εγώ όμως και η ομάδα μου ε, διαφωνούμε με κάποιες ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω να βρεθεί μια συμβεστική λύση ε, αύριο με τον εισηγητή. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη προβλέπω ε, κάποιους επιπλέον ε, διερμηνείς και καμπίνες πολύ σύντομα να προστίθεται σε αυτή την αίθουσα. E Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα ECR υποστηρίζει απόλυτα την ένταξη τη Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αυτή η απόφαση είναι αποκλειστικά υπόθεση τη Ισλανδία σε ένα δημοψήφισμα. Είναι μια μικρή, σταθερή δημοκρατία μέλος ε, του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης η οικονομία της εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αλληλεία. Μετά από το πλήγμα που σημειώθηκε σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, εδώ η Ισλανδία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα των ε, δικών της δυνατοτήτων αλληλεία αν πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική, όσον αφορά την φαλαινοθυρία δεν μου αρέσει ούτε η ταυρομαχία ούτε οι άλλοι είδους ε, ε, τέτοιες εκδηλώσεις και πρέπει να δούμε με την εθνική πολιτισμική παράδοση αν ενταχθεί η Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αν επιμείνει η Ισλανδία να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η πτυχή της ε, φαλαινοθυρίας. Επίσης σε σχέση με την κατάρρευση της ISAF θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημιώσεων και αυτό θα είναι πραγματικά πραγματικά ένα σημαντικό εμπόδιο για να δοθεί υποστήριξη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, στην ε, Βρετανία η 1η Απριλίου είναι η ημέρα των πρωταπριλιάτικων ψεμάτων γίνονται τέτοιου είδους αστεία. Λοιπόν, α, το ότι θα βρίσκεται η Ισλανδία σε πορεία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα πρωταπηλιάτικο αστείο, διότι δείχνει 64% η σφιγμομέτρηση ότι επιθυμούν 64% των Ισλανδών να παραμείνουν ανεξάρτητοι και να μην ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 60% των επιχειρήσεων είναι εναντίον της ένταξης. Άλλοι λένε ότι θα, σε σχέση με την ασφάλεια του ευρώ λέει θα συνεισέφερε και αυτό πρωταπληκτικό αστείο. Ακόμα και σήμερα αρνούνται να αγοράσουν ομόλογα της Πορτογαλίας, της Πορτογαλίας ήδη οι τράπεζες. Και εδώ βλέπουμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί και στην ολέθρια αλλιευτική πολιτική, κοινή αλλιευτική πολιτική. Και βλέπουμε ότι σε σχέση με όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα ακόμα και με τα χρηματοπιστωτικά προβλήματα. Η Ισλανδία όπως ε, και η Μεγάλη Βρετανία καλύτερα να παρέμενε εκτός ευρώ χωρίς πρωταπηλιάτικα αστεία. Ευχαριστώ. Μα είναι 6 Απριλίου σήμερα. Με μπερδέψετε λίγο με την αφορά σας την Πρωταπριλιά. Το έλεγξα. Είμαστε 6 Απριλίου σήμερα. Ναι, μπορείτε να κηρύξετε και την ημέρα αυτή αν θέλετε Πρωταπριλιά. Πολύ ωραία. Mr. President, Κύριε Πρόεδρε, ω συνήθω η συζήτηση εδώ πέρα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και καμία σχέση με τη δημοκρατία. Οι περισσότεροι εδώ πέρα παίρνουν το λόγο σαν να έχει ουσιαστικά ήδη α, ολοκληρωθεί η προσχώρηση τη Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα δημοψηφίσματα δείχνουν ότι οι πολίτε δεν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα 75% των Ισλανδών πολύ σοφά δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο κόμμα της Ισλανδίας υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει πάρα πολύ σημαντική πτώση σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Φαίνεται ότι ενώ οι πολιτικοί ηγέτε θέλουν την προσχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη οι πολίτε τη Ισλανδία προτιμούν να μην είναι κυρίαρχοι. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι εσείς συγχαίρετε τον εαυτό σας για την όλη διαδικασία προσχώρησης. Η ε, κατάρρευση όμως ήδη των κρατών που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκονται στο Ζουρδομανδία της Ευρωζώνης, ουσιαστικά αποτελεί μια πραγματικότητα. Η ε, Ισλανδία και πολλές άλλες χώρες ουσιαστικά πιστεύω θα καταμείνουν τελικά ελεύθερες. ευχαριστώ πολύ, η Ισλανδία είναι φυσικά μια μικρή χώρα με μικρά εισόδα. Παρόλα αυτά όμως είναι ένα μεγάλο έθνος, μεγάλος λαός. Η Ισλανδία έχει δημοκρατικές παραδόσεις εδώ και πολλούς αιώνες. Μια, έναν εντυπωσιακό πολιτισμό και παράδοση. Ένα πολύ καλό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων καλύτερο από τις άλλες χώρες. Φυσικά μπορούμε ιστοδυναικές να συζητούμε για την οικονομική κρίση του 2008. Όμως σε αρκετές χώρες ζήσαμε αυτή την οικονομική κρίση και όχι μόνο στη μικρή Ισλανδία μια μικρή χώρα με 300.000 πολίτες που ιδιαίτερα επλήγει, ιδιαίτερα σκληρά από την κατάρρευση της οικονομίας. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις και στην κρατική διοίκηση και να μην το ξεχνάμε αυτό ότι κάνουμε λόγο για μια νησιωτική χώρα στην, ε, Αρκτική, στην περιοχή του Αρκτικού κύκλου. Και εδώ έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα οι Ισλανδοί όσον αφορά την αλληλεία. Ολόκληρες γενναίες Ισλανδών εξαρτήθηκαν και έζησαν από την αλληλεία. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Κάνουμε λόγο λοιπόν για ένα μικρό έθνος και όχι για ένα τεράστιο έθνος. Η Ισλανδία τούτων λεχθέντων θα πρέπει φυσικά να εξεταστεί ανάλογα με τις ικανότητές της προσένταξη και νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν να πούμε ότι έχουν καλύτερες επιδόσεις Ισλανδοί από ό,τι άλλες χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα θα ήταν για την Νορβηγία σιγά σιγά βαθμιαία να προσεγγίσει αυτή την πορεία προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χαιρετίζουμε αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Η πρόταση ψηφίσματο που έχουμε ενώπιον μας καλύπτει όλα τα βασικά σημεία της έκθεση πρόοδου. Υπάρχουν 33 κεφάλαια και από ό,τι φαίνεται η Ισλανδία κινείται πολύ γρήγορα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση έγινε μια αναφορά στον αφορά την Ειδική Εξεταστική Επιτροπή του Ισλανδικού Κοινοβουλίου στον αφορά την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδοθούν οι ευθύνε και ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να μάθει κάποια διδάγματα από τη λογική προσέγγιση τη Ισλανδία. Θα ήθελα να φερθώ σε δύο ζητήματα. Καταρχά, Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε ευτυχώς να βρούμε μια λύση στο όλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το δημοψήφισμα και πιστεύω ότι από αυτού θα ασχοληθεί και το και το Ισλανδικό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το σκουμπρί, φαίνεται ότι η Ισλανδία έχει πολύ ψηλά ακόμα, πολλές ψηλές ποσοστώσεις ακόμα για τα λιεύματα σκουμπρίου. Πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η προσχώρηση της ε, Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πάτκοτ Γκάλαχερ στο Ρέικιαβικ στις 26 και 27 Απριλίου, όπως σας είπα, θα είναι επικεφαλής της συζήτησης Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, με χαροποιεί το γεγονό ότι η πλειονότητα των Ισλανδών στη δημοσκόπηση που έγινε είπαν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ειλικρινώ, γιατί να θέλουμε να ενταχθούν, τι ακριβώ θα προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διότι έχουν μία χρεοκοπημένη οικονοποιημένα, έχουν τράπεζες που χρεοκόπησαν, το ηφαίστειο έκλεισε τον εναέριο χώρο για εννέα μέρες, δεν ξέρω τι θα κάνουμε άμα να συμβεί κάτι τέτοιο και τώρα απειλούν και τα αποθέματα σκουπριού. Το 2005 η Ισλανδία εκφόρτωσε 367 τόνους ε, ε σκουμπριού του Ατλαντικού. Αυτή τη στιγμή σκοπεύουν να εκφορτώσουν 150.000 τόνους. Τι είδους καλή διαχείριση, βιώσιμη διαχείριση αλίας ε, την αποκαλούμε αυτή. Πάντα περηφανεύονται ότι έχουν βιώσιμη αλία και περιγελούν την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική που αποφαρμόζουμε εμείς. Είναι εγκληματικό. Είναι σχεδόν παράνομη αλία αυτό που κάνουν. Και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να τους προσκαλέσουμε να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα σας πω κάτι που μου είναι ιδιαίτερα προφιλές. Μόνο μία έδρα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Στρασβούργο. Όπως ξέρετε, το σκουμπρί μας μας απασχολεί. Οι τελευταίες ε, διαπραγματεύσεις απέτυχαν. Εδώ και για περισσότερα από 10 χρόνια υπάρχει ε, κλίμακα κατανομής ε, των ποσοτήτων ε, αλίας κουμπρίου. Ζητάει όλο και περισσότερα ποσά η εξαιτία των κλιματικών αλλαγών και της αύξησης της θερμοκρασίας η Ισλανδία. Και έτσι από 2.000 ανέβηκε σε 130.000 τόνους η πέρσι η ποσόστοση που δόθηκε στην Ισλανδία. Πράγμα το οποίο επιβάλλει κυρώ στου δικού μα Δεν μπορούμε να δεχθούμε λοιπόν τέτοιου είδου μονομερεί αποφάσει να λαμβάνουμε. Θέλουμε να ρυθμιστεί το συντομότερο δυνατό το θέμα αυτό που αποκαλεί μια διένεξη. Η Ισλανδία θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κοινή ελευθερική μας πολιτική και όχι το αντίθετο. Παίζει επικίνδυνο παιχνίδι η Ισλανδία, διότι με σε επιβάλλει απαράδεκτου όρου Θα πρέπει να κάνει η πολιτική πιο ρεαλιστική. Τελικά κανένας δεν θα ήθελε υπεραλίευση και την θέση εν κινδύνο των αποθεμάτων σκουμπριού. Θα ήθελα να επιδείξει πνεύμα ευθύνη και ευελιξία στην διαπραγματεύση Ισλανδία και περισσότερη διαφάνεια στι συζητήσει. Σα ευχαριστώ. τέσσερι ομιλητέ. Πρώτο ο Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ισλανδία διότι πλέον υποψήφια χώρα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προετοιμασία της Ισλανδίας είναι σε καλό δρόμο και συνάδει και με το χρονοδιάγραμμα. Α μην λησμονούμε όμως ότι οι προποθέσει ένταξης είναι και η δέσμευση τη κυβέρνηση, αλλά και του λαού. Οι κατάλληλες πληροφορίες λοιπόν προς την κοινή γνώμη είναι στοιχείο κλειδί για την αποτελεσματική ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπειρία της Πολωνίας καταδεικνύει ότι δεν αρκούν μόνο οι εκστρατείε ε, τη κυβέρνηση και των μέσων μαζική ενημέρωση, αλλά και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και η διεθνή συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι η Ιρλανδία έκανε πάρα πολλά πράγματα για την ανάπτυξη, για την παιδεία και τα πλαίσια της στρατηγικής της ε, Λισαβένας. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει και ε, λάβει και διάφορα μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Πιστεύω ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας ε, θα είναι επωφελής για όλους. Θα, Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να έχει πρόσβαση στην ε, περιοχή αυτή της Αρκτικής που είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως θα λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές. Πιστεύω λοιπόν ότι ο διάλογος ε, θα πρέπει να εντεθεί. Η σύστασή μου λοιπόν είναι για τους Ισλανδούς που ελπίζει τελικά αποτελέσματα ε, θετικά να δοθεί το πράσινο φως. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συγχαρούμε αυτούς το γεγονό ότι η Ισλανδία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί απόδειξη του γεγονότο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιο κύρο ε, και η ασφάλεια, η εφημερία και ε, η ανάπτυξη που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιτυχία και γι' αυτό και ακριβώ μια χώρα σαν την Ισλανδία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια και η οικονομική κρίση διαδραματίζει το ρόλο τη ε, στην απόφασή του αυτού. Η ένταξη βέβαια τη Ισλανδία δεν θα πρέπει να γίνει αυτομάτω. Θα πρέπει να δούμε τι επιπρόσθετο όφελο μπορεί μπορεί να προσδώσει η Ισλανδία σε εμά. Ήδη μεγάλο τμήμα της Ισλανδικής νομοθεσίας είναι συμμορφούμενοι προς την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν και στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Η Ισλανδία είναι μια αγαπητή και πλούσια χώρα και ελπίζω ότι θα βεβαιωθούμε ότι πληρούνται όλα τα κλητήρια για την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση για την ένταξη της Ισλανδίας. Ευχαριστώ Η έκθεση πρόοδου για την Ισλανδία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από διάφορε πτυχέ. Είναι μια δημοκρατία, μια χώρα που πληρεί όλε τι προποθέσει από πλευρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μέλος της ελεύθερης ζώνης εμπορίου, της ΕΖΕΣ και σε πολλές περιπτώσεις ε, συμμορφούνται με το κοινοτικό κεκτημένο. Σε αντίθεση με άλλες χώρες λοιπόν έχει το προβάδισμα. Παρά το γεγονός ότι η Ισλανδία έχει μια καλά λειτουργούσα οικονομία αγοράς και είναι ενταγμένοι στο χρηματοοικονομικό τομέα και υπάρχουν στοιχεία στο τραπεζικό σύστημα που μας ανησυχούν. Η κατάστασή της βελτιώνονται, αλλά ε, υπάρχουν ε, σημαντικά ποσοστά πληθωρισμού και η αυξανόμενη ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η Ισλανδία θα πρέπει να ενισχύσει την ανεξαρτησία του δικαστικού της ε, ε, συστήματος. Έχει κάνει αρκετή πρόοδο σε θέματα παιδείας ε, και είναι αρκετά ανταγωνιστική με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συμμετέχουν σε πολλά προγράμματα όπως το Erasmus Mundus και νομίζω ότι πρόκειται για μια σταθερή δημοκρατία με σταθερούς θεσμικούς ε, θεσμούς. Thank you very much, Mr. President, members. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε εξαιρετικά μέλη του Κοινοβουλίου. Η σημερινή συζήτηση ήταν παραγωγική και εντόπισε τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ισλανδία για να έχουμε ε, θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις. Όπως αναγνωρίζετε στο ψήφισμα το οποίο ε, συζητήσαμε και την έκθεση πρώτη προηγούμενου Νοεμβρίου, η Ισλανδία βρίσκεται σε ε, προχωρημένο στάδιο όσον αφορά τα κριτήρια που πληρεί, αλλά θα πρέπει σε κάποια συγκεκριμένα θέματα να υπάρξει περαιτέρω πρόεδρος. Κάποιοι από εσά ανέφεραν το θέμα του σκουμπριού. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα θέματα αφορούν κυρίως την διαχείριση των αποθεμάτων στον ε, ε, βορειοανατολικό, συγγνώμη, Ατλαντικό, σε σχέση με όλες τις παράκτιες χώρες, μας απογοητεύει η έλλειψη πρόοδου που διαπιστώσαμε επί αυτού του θέματος στις τελευταίες διαβουλεύσεις. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές απόψεων, κυρίως μεταξύ της ε, Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και των νησιών Φεροέ και της Ισλανδίας από την άλλη όσον αφορά το αντίστοιχο μερίδιο του καθενός η αηφορία και η βιωσιμότητα αυτού του πόρου είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αλληλευτική μας βιομηχανία και θα συνεχίσουμε εμείς να ανοιχνεύουμε όλους τους δρόμους ώστε να μπορέσουμε να δούμε ισοσκελισμένη λύση για όλες τις περιοχές, της ε, τις χώρες περιοχής αυτές. Η Ισλανδία, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή μπαίνει σε ένα αποφασιστική συζημίας στάδιο. Είναι θέμα δικής της αποφασιστικότητας το να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις και εάν δεν υπάρξει και υποστήριξη των πολιτών της δεν θα μπορέσει η Ισλανδία να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σαφώς ε, παρουσιάστηκαν αρκετά ζητήματα και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα προσπαθήσει να λάβει υπόψη όλες αυτές τις πτυχές. Θα ήθελα να πω ότι βάσει του προγράμματός μας εγώ θα είμαι παρόν στη συνεδρίαση που θα γίνει στα τέλη Απριλίου στο Κοινό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας και σε εκείνη την περίπτωση θα μπορέσουμε να έχουμε και πιο διεξοδικές πληροφορίες από πλευράς των Ισλανδικών αρχών για κάποια ζητήματα. Βεβαίως όσον αφορά τη γεωργία και την αλληλεία ή το θέμα του iSave, Υπήρξαν προβλήματα, αλλά είμαι βέβαιη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα με τη δέουσα διαφάνεια και σαφώς όσο θα προχωρούν οι διαπραγματεύσεις ένταξης θα ε, ενημερώνει και τους ευρωβουλευτές αναλόγως. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι με ευχαριστή ιδιαίτερα το γεγονό ότι κανεί από όσου παρενέβησαν στη συζήτηση δεν αμφισβήτησε το γεγονό ότι η Ισλανδία έχει μια πολιτική κουλτούρα και ένα δημοκρατικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με αγαστό τρόπο. Γι' αυτό και ακριβώς είμαστε βέβαιοι όλοι ότι οι Ισλανδοί θα λάβουν μία απόφαση ε,